Ladies and gentlemen, welcome and let us continue by item number 10. Ας συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι με το θέμα 10 που είναι η παρουσίαση της μελέτης ε, τεχνητή νοημοσύνη και αστικό δίκαιο κανόνες περιευθύνης ε, για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και η μελέτη αυτή εκπονήθηκε μετά από αίτημα της Επιτροπής μας. Αναλύουμε τις εθνικές νομοθεσίες σε σχέση με τη χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών όπου προαπαιτείται ε, καταγραφή, εγγραφή σε μητρώα και πιστοποίηση και υποχρεωτική ασφάλιση. Τέλος, με βάση την διαχείριση κινδύνου, η έκθεση μιλά για την εξέλιξη, μελλοντική εξέλιξη του ζητήματος. Ο κύριος Ανδρέα Μπερτολίνη θα κάνει την παρουσίαση, ο οποίος εργάζεται στην Σκόλα Σουπεριόρε Σαντάνα στην Πίζα και Επίσης ασχολείται με το ιδιωτικό δίκαιο ε, με βάση τα δεδομένα ε, ως προς την εξέλιξη του ζητήματος, δύναμη του ιδιωτικού δικαίου. Αυτή η μελέτη έχει σαν στόχο την αναγνώριση των ζητημάτων που σχετίζονται με την πιστοποίηση των μη επανδρομένων αεροσκαφών για ιδιωτική χρήση, καθώς και θέμα ευθύνης και ασφάλισης. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε και μετά θα μιλήσω για τα κριτήρια ταξινόμησης των μη επανδρομένων αεροσκαφών όπως ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα. Μετά θα μιλήσω για τους κανόνες περί και την ασφάλιση. Σε σχέση με τους στόχους, καταρχήν, η μελέτη έχει στόχο να δώσει μία συνολική εικόνα των ορισμών και ταξινομήσεων μέσα στα πλαίσια των κανόνων περιευθύνης και στη συνέχεια προβαίνει σε συστάσεις με βάση βεβαίως τον νόμο περί ευθύνης, την ασφάλιση και την διαχείριση κινδύνου. Και στα πλαίσια αυτά δίνει ένα γενικό ορισμό, ε, μια συνολική εικόνα, με συγχωρείτε, των ορισμών που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Γιατί έχει μεγάλη σημασία, έχει τόση σημασία, ποιοι είναι οι ορισμοί που χρησιμοποιούμε τους χρησιμοποιούμε για να γίνει σωστή ταξινόμηση, γιατί υπάρχει διαφορετική ταξινόμηση των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ας δούμε πώς έχει η ευρωπαϊκή ρύθμιση. Υπάρχει ο πρόσφατος κανονισμός του 2018 σε σχέση με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τον επιμερισμό ευθυνών, όπου μιλάμε για οποιοδήποτε όχημα αέρος το οποίο μπορεί κανείς να χειριστεί, ε, να, προβεί μάλλον σε τηλεχειρισμό αυτών των αεροσκαφών χωρίς να υπάρχει πιλότος επί του σκάφους. Φυσικά εδώ υπάρχει ένα συνολικός βαθμός ε, κινδύνου Επίσης υπάρχει ένα συνολικός ε, βαθμός κινδύνου ένα συνεκτικός βαθμός κινδύνου, δηλαδή δεν πρόκειται για μία διάκριση που βασίζεται στον όγκο όπως ισχύει σε άλλα κράτη-μέλη ή στις ΗΠΑ, αλλά άλλες πτυχές λαμβάνονται υπόψη που έχουν σημασία. Δηλαδή οι άλλοι κίνδυνοι που ενέχονται ως προς την ιδιωτικότητα και τα άλλα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να έχει αισθητήρε το μη επανδρομένο αεροσκάφος, για παράδειγμα. Άρα ορίζονται κατά διαφορετικούς τρόπους και έχετε έναν πίνακα που σας δίνει όλα τα κριτήρια ταξινόμησης και ορισμών. Δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά τα περισσότερα κράτη-μέλη τα ταξινομούν ανάλογα με το βάρος τους. Όμως, ο κανόνας που ισχύει πλέον με βάση τον κανονισμό λαμβάνει υπόψη και άλλα κριτήρια. Διαφορετικά στις ΗΠΑ μιλάμε για ε, οχήματα αέρος τα οποία χειρίζεται κανείς εξ αποστάσεως χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία μέσα στο ίδιο το όχημα αέρος. Και δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο τους ε, τηλεχειρισμούς ή τους αυτόνομους ε, χειρισμούς. Επίσης, ε, οι ΙΠΑ λαμβάνουν υπόψη για την ταξινόμηση το βάρος και την λειτουργία. Αυτά είναι τα δύο κριτήρια ταξινόμησης των μη επανδρομένων αεροσκαφών στις ίπα και επίσης ποιος, ε, γιατί χρησιμοποιούνται, ποιος είναι ο πότερος στόχος αναψυχής, ε, εμπίπτει στο ιδιωτικό δίκαιο ή στο δημόσιο. Τα κράτη-μέλη, όπως σας είπα, πρωταρχικά ταξινομούν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ανάλογα με το βάρος τους, αλλά αυτό δεν είναι και το μοναδικό κριτήριο η πτυχή, γιατί σας είπα πέραν αυτών των κατηγοριών μπορούν να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια για να ταξινομηθούν. Ουσιαστικά βασιζόμενοι στον ευρωπαϊκό κανονισμό, μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο λογική η κατηγοριοποίηση. Υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή σε, στα ευρωπαϊκά κείμενα σε σχέση με α, επιμέρους εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. ταξινόμηση του κινδύνου στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές που ουσιαστικά υπολογίζουν και αξιολογούν ε, τον κίνδυνο και τις ε, απαιτήσει όσον αφορά την πιστοποίηση. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν διαφορετικές ε, παράμετροι που οδηγούν σε μια συγκεκριμένη ταξινόμηση και βεβαίως όλες αυτές οι παράμετροι οδηγούν σε κατηγορίες ασφάλισης και τις καλύτερες προϋποθέσεις και κανόνες που αφορούν την ευθύνη. Αυτό βέβαια δεν εξαρτάται άμεσα από την αξιολόγηση του κινδύνου. Η εμπορική και η μη εμπορική χρήση των ε, drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών, που θα μας οδηγήσουν πολλές φορές σε διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά την ασφάλισή τους. Θα επανέλθω σε αυτό. Όσον αφορά τους κανόνες για περί η ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει σε μεγάλο βαθμό το θέμα της αξιολόγησης του κινδύνου. Αυτό βεβαίως εδώ και βασίζομαι στον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία που ουσιαστικά ισχύει εδώ για όλα τα υπτάμενα οχήματα πρόκειται για την οδηγία του 2004 που αφορά την ασφάλιση, τις προϋποθέσεις για την ασφάλιση των ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών. Αυτό βεβαίως ισχύει για να μπορέσει να καθοριστεί η ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. Ο κανονισμός δεν αφορά συγκεκριμένα θέματα ευθύνης. Γι' αυτό και παραμένει εδώ ένα μεγάλο κενό όσον αφορά τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι εθνικές νομοθεσίες. Το θέμα είναι ποιος είναι ο χρήστης. Αν είναι φυσικό πρόσωπο. Και αυτό βεβαίως είναι λογικό και ενδεχομένω μπορεί να μας οδηγήσει στην προτιμονόμενη, αν θέλετε, λύση σε πολλά κράτη-μέλη, σε πολλές εθνικές ε, νομοθεσίες. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί, λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί της πολιτικής αεροπορίας. Και εδώ βεβαίως πολλές φορές δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τους ίδιους κανόνες ε, στα μη επανδρομένα αεροσκάφη που εφαρμόζονται στα παραδοσιακά αεροσκάφη. Γι' αυτό και πολλά μέλη έχουν αποκλείσει κάποιους από τους κανόνες που ισχύουν για την πολιτική αεροπορία. Το θέμα λοιπόν της ευθύνης. Πώς μπορεί δηλαδή να αποδειχθεί ποιος είναι υπεύθυνο η χρήση των κανόνων ευθύνης που προϋποθέτουν ένα φυσικό πρόσωπο χειριστή και βεβαίως την υποχρεωτική ασφάλιση αυτών των ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και εδώ θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των ε, εμπορικών και των μη εμπορικών χρήσεων και πτήσεων. Βλέπετε εδώ σε αυτό το χάρτη με πορτοκαλί χρώμα τις χώρες που έχουν επιλέξει ε, συγκεκριμένους κανόνες περί ευθύνης και με πράσινο χρώμα, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, την Ιρλανδία και την ε, Τσεχία, που εδώ έχουν επιλέξει την ευθύνη του χειριστή. Οι διαφορές εδώ είναι πολύ σημαντικές, θεωρητικά τουλάχιστον, αλλά και στην πράξη διότι διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ πιο απλή η κατάσταση όταν ισχύουν οι σαφείς κανόνες περί σε περίπτωση παραδείγματο χάρη ατυχήματος. Η λειτουργία του μη επανδρομένου αεροσκάφους, ο χρήστης αυτού, ο χειριστής αυτού και βεβαίως η παράμετροι που διέπουν αυτή τη λειτουργία. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε, ιδιαίτερα σε εμπορικές πτήσεις, να υπάρχουν περισσότεροι χειριστές. Συνήθως ένα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρεμένο αεροσκάφος ε, έχει ένα χειριστή. Αυτό όμως δεν είναι ε, κάτι που ισχύει πάντοτε. Στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες για την πιστοποίηση και κάθε φορά υπάρχει η νομοθεσία των πολιτιών. Οι ρυθμίσεις, οι κανονισμοί και η ευθύνη ουσιαστικά απορρέουν από την ύπαρξη ενός φυσικού προσώπου, του χρήστη. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει ευρύτερο φάσμα από αυτό των πολιτιών. Και για μένα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα περιπτώσεων που δεν καλύπτονται από την νομοθεσία αυτή. Προσπαθώ να σας δώσω μια γενικότερη εικόνα του τι ισχύει και ολοκληρώνοντας θα σας πω ότι για την αξιολόγηση του κινδύνου το θέμα του εντοπισμού των ευθυνών και το θέμα της ασφάλισης που απορρέει από αυτά είναι κάτι που θα πρέπει να οριστεί σίγουρα ορίζοντας σαν κεντρικό πρόσωπο τον χειριστή και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ευθύνη απορρέει κυρίως από αυτό το κεντρικό πρόσωπο τον χειριστή. Και βεβαίως διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες ε, εθνικές νομοθεσίες στην Ευρώπη δεν ε, ανταποκρίνονται σε αυτήν την ε, βασική αρχή, καθότι καθορίζουν διάφορες ε, ε, κατακαιρματισμένες ε, ευθύνες. Διαπιστώνουμε επίσης ότι οι εθνικές νομοθεσίες είναι εντελώς διαφορετικέ. Θα προσπαθήσω την ίδια ώρα να διαπιστώσω ότι η τεχνολογία ορίζει σε μεγάλο βαθμό ε, τους κανόνες περί ευθύνης. Οι κατασκευαστέ, παραδείγματο χάρη, στα διάφορα κράτη-μέλη στην Ευρώπη, μπορεί να έχουν υιοθετήσει και επιλέξει τελείως διαφορετικές νομοθεσίες, κάτι το οποίο έχει καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την νομοθεσία τους. Αυτό λοιπόν το επιπλέον στοιχείο σίγουρα θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια πιο ομοιογενή ευρωπαϊκή προσέγγιση από αυτήν που έχουν επιλέξει τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ποια είναι τα συμπεράσματά μου και οι συστάσεις μου. Όσον αφορά την ασφάλιση των μη επανδρομένων αεροσκαφών, θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση του κινδύνου και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βασιστούμε στον ε, κανονισμό του 2018. Θα πρέπει αυτό να θεωρηθεί ότι είναι η πιο κατάλληλη νομική βάση. Παρόλα αυτά, όλα τα μη ε, επανδρομένα αεροσκάφη θα πρέπει να έχουν υποχρέωση καταγραφής σε Μητρώα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και ποιος είναι ο χειριστής. Αυτό σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών είναι κάτι που ε, έχει περάσει στην νομοθεσία. Οποιοδήποτε μη εμπαδρομένο αεροσκάφος που ξεπερνάει τα 250 γραμμάρια θα πρέπει να καταχωρηθεί σε μητρό. Ακόμα και τα πιο μικρά ε, μη επανδρομένα αεροσκάφη καταγράφονται λοιπόν σε μητρό σε επίπεδο πολιτιών. Ολοκληρώνω λοιπόν, και αυτό είναι και το συμπέρασμά μου, Σίγουρα θα πρέπει να περάσουμε στις ε, ε, προδιαγραφές περί ευθυνών βασιζόμενοι σε αντικειμενικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες τεχνολογίες σίγουρα οδηγούν σε εξέλιξη των ε, νομοθεσιών και θα πρέπει να υιοθετήσουμε και μία προσέγγιση one-stop shop σε όλη την Ευρώπη. Όποιος και να είναι ο κατασκευαστής, όποιος και να είναι ο πιλότος, όποιος και να είναι ο χειριστής ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους, δεν θα πρέπει να υπάρχει δυσκολία εντοπισμού όσον αφορά την προσφυγή σε περίπτωση ατυχήματος και θα πρέπει εξάντε να υπάρχει καθαρός εντοπισμός, σαφή κριτήρια όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου και να μπορούμε να προσφύγουμε είτε κατά του πιλότου, είτε κατά του κατασκευαστή, κατά του χειριστή. Θα πρέπει το θύμα επίσης να μπορεί να εντοπίζεται με σαφέστατο τρόπο και σαφείς κανόνες ε, από την νομοθεσία. Όσον αφορά τη χρήση ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους. Σίγουρα ο χειριστής είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπορεί να εντοπιστεί με σαφέστατο τρόπο. Εάν κοιτάξουμε τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ανατρέξουμε στον ιδιοκτήτη και όχι στο χειριστή του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ασφάλιση κατά τρίτου για κάθε είδους μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε εκτελούν μη εμπορικές είτε εκτελούν εμπορικές ε, πτήσεις και αυτό θα πρέπει να καλύπτει ενδεχομένως και τα μικρότερα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να παραμείνουν όλες αυτές οι προδιαγραφές που αφορούν την ασφάλιση στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι και ο κανονισμός του 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει όλες τις κατηγορίες των μη επανδρομένων αεροσκαφών, όλα τα μεγέθη και τις δυνατότητες ε, να εμπεριέχονται κάμερες ή άλλοι μηχανισμοί. Οι προϋποθέσεις λοιπόν για την ασφάλιση όπως είπα και προηγουμένως θα πρέπει να καλύπτουν ε, με ασφάλιση κατά τρίτον όλες τις κατηγορίες των μη επανδρομένων αεροσκαφών, γιατί ακόμα και οι μη εμπορικές πτήσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, ε, να παραβιάζουν παραδείγματος χάρη την ιδιωτικότητα και θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός της υπάρχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ο κανονισμός του 2018 καθώς και ο κανονισμός για ασφάλιση του 2004, καθώς δεν υπάρχει κανένα συντονισμός μεταξύ των δύο αυτών κειμένων. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις προς τα θύματα, Έχει αναφερθεί η ανάγκη για να υπάρξει ένα ταμείο αποζημιώσεων και την κάλυψη των ε, περιπτώσεων ατυχημάτων. Ένα ποσοστό θα πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό το ταμείο δεν ανακαλύπτονται οι τυχόν ε, ζημιές για μικρότερα μη επανδρομένα αεροσκάφη που πολλές φορές ε, δεν, υποχρε... δεν είναι <clears throat> υποχρεωτική η ασφάλισή τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι η εναρμόνιση της νομοθεσίας είναι κάτι το απαραίτητο, όχι μόνο γιατί θα δημιουργηθεί αυτή η υποχρέωση για ασφάλιση για όλα τα μία παντρωμένα αεροσκάφη στην Ευρώπη και θα καλύψει την, τις διαφορετικές νομοθεσίες που σήμερα υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη, καθώς και την διαφορετική νομοθεσία που οφείλεται σε διαφορετική τεχνολογία. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει περισσότερος κατακαιρματισμός πέραν αυτού που σήμερα προκύπτει από τις διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος να θέσει κάποιο ερώτημα, ιδιαίτερη κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Αντρέα για την παρουσίαση. Έχω μπερδευτεί λίγο κάνεις λόγο για μια νέα ταξινόμηση το 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη-μέλη και δεν υπάρχει διαφορά ε, εκτός ε, μόνο από το γενικό βαθμό κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αλλάξουν τους κανόνες επειδή υπάρχει νέα ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ευρωπαϊκής ταξινόμησης και αυτή των κρατών μελών. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και η δεύτερη ερώτηση. Υπέρ της καταχώρησης όλων των ε, μη παντρωμένων ε, ε, σκαφών έχω εγγόνια που θέλουν drones για τα Χριστούγεννα. Αν είναι δηλαδή παιχνίδι, θα πρέπει να το κατα γράψω και άλλη μια ερώτηση που αφορά την ε, ποινική ευθύνη. Ο παραγός είναι υπεύθυνο σύμφωνα με την νομοθεσία για τα λατώματα. Από ό,τι κατάλαβα και ο χειριστής θα είναι υπεύθυνο για παραβίαση ιδιωτικότητας. Είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει βλάβη λόγω ελαττώματος ή παραβίασης ιδιωτικότητας. Πώς το ορίζεις αυτό ή κάτι δεν κατάλαβα καλά μάλλον. Ναι, θα προσπαθήσω. Για την καταγραφή και τις σχετικές προϋποθέσεις στις Ηνωμένες κάθε drone πάνω από 250 γραμμάρια πρέπει να είναι καταγεγραμμένο. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το βαθμό ή ε, να εξαιρέσουμε τα παιχνίδια drones ή που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς σκοπούς και πολύ μικρού μεγέθους. Οι προποθέσει μπορούν ε, για την καταγραφή πρέπει να διαχειριστούν πολύ απλά. Κάτι τέτοιο στη ΣΥΠΑ μπορεί να συμβεί στο ίντερνετ, online. Κάποιο αγοράζει π.χ. ένα παιχνίδι το οποίο ζυγίζει πάνω από 250 γραμμάρια και είναι πολύ εύκολο κανεί να το καταγράψει. Ε, online. Όμως ε, σε μεγαλύτερα μεγέθη είναι πιο περίπλοκη, στις διαδικασίες. Θεωρώ ότι αυτό παρέχει μια βεβαιότητα σε όλο το μηχανισμό. Το πρώτο ερώτημα είχε να κάνει με για τα κράτη-μέλη, ναι τη σχέση. Λοιπόν, είναι εφαρμοστέ ο κανονισμό, είναι ο κανονισμό στα κράτη-μέλη. Ο συντονισμό μεταξύ ε, του κανονισμού και των μεμονωμένων κρατών μελών είναι περίπλοκο. Θα πρέπει να δούμε τι ε, ε, λεπτομέρειε για το καθε κρατη κράτο-μέλο. Ε, είναι ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά αν η, υπάρχει σύγκρουση, υπερισχύει ο κανονισμός, ο οποίο υπερέχει έναντι τη εθνική νομοθεσία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι το μέγεθος του μη πατρωμένου σκάφους. Διερευνήθηκαν οι μελέτες που είχαν γίνει ε, τα προηγούμενα χρόνια από την Επιτροπή για τους κινδύνου που έχει τον τρόλο, όχι μόνο του βάρους, αλλά και της ανέργειας που έχει του ύψους στο οποίο πετάει και επίση τα διάφορα θέματα τα οποία αγγίζει. Λάβανε υπόψη λοιπόν όλες τις πτυχές, όλες τις πολύπλοκες πτυχές. Τώρα πώς αυτό ε, συγκρούεται με τι εθνικέ νομοθεσίε, θα πρέπει να το δούμε μεμονωμένα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μπορεί να επηρεαστεί η εθνική νομοθεσία εφόσον ο κανονισμό είναι άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την ποινική ευθύνη, υπάρχουν διαφορετικά είδη κινδύνων. Και η βασική ανησυχία είναι να εντοπίσουμε ποιος είναι υπεύθυνο έναντι του θύματος, ώστε το θύμα να μην ε, βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ξέρει αν έχει να κάνει το ατύχημα με κάποιο ελάττωμα που υπήρχε ή με κάτι άλλο ή με το χειρισμό π.χ. του ντρόν. Θα πρέπει να υπάρχει προστασία της σωματικής κυριότητας σε περίπτωση ε, πτώσης ε, του ντρόν και επίσης υπάρχουν και θέματα Προστασία προσωπικών δεδομένων κτλ. Υπάρχει κερματισμό λοιπόν. Και εξ αυτού μειώνονται οι δυνατότητες ε, αποζημίωσης για τα θύματα. Άρα αυτό πρέπει να γίνει, να εντοπιστούμε, να εντοπίσουμε μάλλον αντικειμενικά ποιος είναι υπεύθυνο και να υπάρχει μια σχετική μορφία μεταξύ κρατών μελών και κυρίως όταν θεωρείται υπεύθυνο ο χειριστής. Θεωρώ ότι αυτή η λύση είναι πολύ λογική. Αν συνδυαστεί με την προσέγγιση του One Stop Shop, τότε θα μπορεί το θύμα να κάνει προσφυγές για τις μεμονωμένες ε, βλάβες που μπορεί να έχει υποστεί και έτσι να μειωθεί και το κόστος της δικαστικής διαδικασίας. Γιατί αν το κόστος είναι υψηλό μπορεί να, είναι να αποφέρονται τα θύματα στο να ζητήσουν αποζημίωση. Ο λόγος στην Επιτροπή για σχόλια. Yes. Uh, hello, I'm uh, Γεια σας, είμαι η Κλάρα Μαρτίνες. Είμαι υπεύθυνη στην ε, είμαι υπεύθυνη για αυτή την ε, οδηγία περιπινικής ευθύνης η οποία ως ένα βαθμό είναι πολύ σχετική ως προς τον ορισμό της ευθύνης των κατασκευαστών. Η πρόκληση όμως είναι πώς θα αποδείξουμε ότι όταν υπάρχουν ελαττώματα ή τραύματα που έχουν προκληθεί από τα drones οφείλονται σε ελαττώματα ή σε λάθος του χειριστή. Ωστόσο, θεωρούμε ότι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο η ύπαρξη αυτής της οδηγίας, ακόμα και αν είναι του 85, δίνει τη δυνατότητα για αποσμίωση στα θύματα. Μελλοντικά πλαίσια ποινική ευθύνη συζητώνται επί του παρόντο σε ομάδε εμπειρογνωμόνων. Υπάρχουν δύο ομάδε εμπειρογνωμόνων που ε, ασχολούνται με ποινική ευθύνη για προϊόντα, προϊόντων όπω τα drones και υπάρχουν δραστηριότητε από πλευρά τη Επιτροπής για την έκδοση εκθέσεων και για να δίνει προσανατολισμό για την ε, ασφάλεια που έχουν να κάνουν με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Επίσης γίνεται και μια αξιολόγηση για τις ε, συνεχιζόμενες αυτές ε, συζητήσεις στο επίπεδο της ποινική ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you Κύριε Κάβαντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση προς τον ε, προσκεκλημένο μας. Πώς βλέπετε την κατανομή των ευθυνών, την ισορροπία των ευθυνών. Προτείνατε κάτι για τους κατασκευαστές. Έχω την εντύπωση ότι προς τα εκεί κατευθύνονται και η Επιτροπή, αλλά και το θέμα του χειριστή, του πιλότου. Κάποιος ο οποίος χειρίζεται με επικίνδυνο τρόπο ένα τέτοιο αεροσκάφος μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντικές ανητικές συνέπειες. Πώς λοιπόν βλέπετε την κατανομή αυτών των ευθυνών. Να ξεκαθαρίσουμε, ο χειριστής δεν είναι ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής του ντρόν βεβαίως και μπορεί να έχει ένα τμήμα της ευθύνης. Το θέμα όμως του χειριστή και του χειριστή για εμπορικούς ε, σκοπούς είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να μας απασχολήσει όταν μιλάμε για την ευθύνη. Πρέπει να εντοπίσουμε λοιπόν καταρχήν τον κύριο υπεύθυνο και μετά να υπάρχουν ε, τα διάφορα επίπεδα ευθυνών, αν θέλετε. Ο χειριστής, υπεύθυνος για οτιδήποτε εξαρτάται και απορρέει από το, τη χρήση του ντρόν και κατόπιν τα άλλα επίπεδα και οι διαφορετικές ευθύνες. Και νομίζω ότι υπάρχουν εμπειρογνώμονες όχι μόνο στην Επιτροπή που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Εγώ δεν ξέρω υποθέσεις που ήδη αν, αν θέλετε εμπλέκονται μη επανδρομένα αεροσκάφη. Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικός και ο ε, ρόλος του πιλότου. Πρέπει να έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες ε, όσον αφορά την ασφάλεια των πτήσεων για μεγαλύτερα drones. Το θέμα των αποζημιώσεων των θυμάτων πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει καταρχήν ο κύριος υπεύθυνο να είναι ο χειριστής και κατόπιν ο, το θύμα θα πρέπει να μπορεί να απευθυνθεί για αποζημίωση καταρχήν στον χρήστη, στον χειριστή και αν υπάρχει πρόβλημα σχεδιασμού ε, του μη επανδρομένου αεροσκάφους να μπορεί να απευθυνθεί κατά δεύτερο λόγο και στον ε, κατασκευαστή. Να υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία με δύο στάδια. Καταρχήν εντοπίζουμε τον ε, κύρια υπεύθυνο τον χειριστή και κατόπιν ο κατασκευαστής. Η πιστοποίηση, η άδεια χρήσης ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους, ε, ο πιλότος επίσης ότι έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για να χειριστεί ένα τέτοιο αεροσκάφος. Και όπως ε, ακριβώς ορίζει η Βρετανική νομοθεσία, δεν νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να επιλέξουμε ως κύριο υπεύθυνο τον πιλότο. Τι εννοείται αυτόν που εκμεταλλεύεται το μη επανδρομένο αεροσκάφος, γιατί αν ο κατασκευαστής, παραδείγματος χάρη, είναι ε, Κινέζος και κάποιος αγοράσει και πουλήσει αυτό το συγκεκριμένο, αν θέλετε, μη επανδρομένο αεροσκάφος. Ποιος είναι υπεύθυνο. Γιατί ένα πολύ καλό μη επανδρεμένο αεροσκάφος, όσο και καλή να είναι η κατασκευή του και ασφαλής, μπορεί να προκαλέσει καταστροφές, εάν ο χειριστής είναι επικίνδυνος. Σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, το θέμα είναι σχετικό, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ο ετών αποζημίωση. Αν ε, έχει εμπορική χρήση το μη επανδρομένο αεροσκάφος, τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά. Εγώ, ε, αν έχω ένα πρόβλημα με μία αεροπορική εταιρεία ποτέ δεν θα προβάλλω αξιώσεις ή δεν θα κάνω αγωγή κατά του πιλότου, αλλά κατά της αεροπορικής εταιρείας. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Για να είναι υπεύθυνο ο πιλότος υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Υπάρχει βεβαίως, ε, υπάρχουν και ποινικά αδικήματα. Μπορούν να υπάρχουν και διοικητικοί κανόνες που επιβάλλουν συγκεκριμένες χρηματικές κυρώσεις κατά του πιλότου έτσι ώστε να ε, μπορεί να ανταποκρίνεται υπεύθυνα. Θα πρέπει να δούμε τους κανόνες περί στα πλαίσια του αστικού δικαίου και αποζημίωση προς το θύμα. Αν ε, το σύστημα είναι πιο κατακαιρματισμένο με πολλούς υπεύθυνου, τότε το θύμα θα πρέπει να επιλέξει ποιον, ε, σε ποιον θα κάνει αγωγή, δηλαδή τον επιχειρηματία, τον πιλότο, αυτόν που μεταχειρίζεται, χειρίζεται το αεροσκάφος. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το εμπλεκόμενο μέρος, ένας ε, φορέας, ε, εμπορικός φορέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος σε αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και τις διασαφηνήσεις σας, αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε δυστυχώς για να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη. Με την ημερήσια διάταξη σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Συνεχίζουμε με το θέμα υπαριθμών 11 θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Μωρέν Σαρτιέ που μέχρι το τέλος του 2018 ήταν η συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των παιδιών. Η κυρία Μωρέν Σάρτιε θα μας παρουσιάσει την έκθεση δράσης και συστάσεις κατά τη διάρκεια της εντολής της από τον Ιανουάριο του 17 μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου του 18. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, κυρία Μωρέν Σαρτιέ μετέτρεψε το ρόλο του διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σε θέματα που άπτονται τις απαγωγές απογωνής σε ε, διεθνές πλαίσιο. Και αυτό αφορά την, ε, τις διασυνοριακές απαγωγές. Δούλεψε λοιπόν άοκνα για να μπορέσει να αποτιμήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά και τις οικογένειες και μέσα στα πλαίσια και της νέας εντολής, τον Απρίλιο του 2018 από το Προεδρείο, ε, συντόνισε τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να φτάσει σε ένα ε, σημείο, να εστιάσει την προσοχή της σε ένα σημείο ή σε συγκεκριμένα σημεία εντός Κοινοβουλίου και εκτός. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κυρία Μωρέν Σαρτιέ. Και επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Κοράτσα Μπίλτ που ανέλαβε το ρόλο της συντονίστριας από τον Ιανουάριο. Δεν θα μπορέσει όμως να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση γιατί βρίσκεται στην Ουκρανία ως παρατηρήτρια των εκλογών, της εκλογικής διαδικασίας, αλλά σας στέλνει θερμούς χαιρετισμούς. Η κυρία Μωρέν Σαρτιέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, που με καλωσορίζετε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Πρέπει να το κάνω ενώπιον της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων πριν υποβάλω την έκθεση αυτή στο Προεδρείο. Αυτή είναι η τακτική διαδικασία, αλλά είναι και μεγάλη μου χαρά να το κάνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε χρόνο και να συζητήσουμε αυτή την εργασία. Πράγματι, ανέλαβα την ευθύνη την συντονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Ιανουάριο 17 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μέρετ Μαγκίνες και την Άννα Μαρία Κορατσαμπίλτ. Η Μέρετ Μαγκίνες ήταν προκάτοχος αυτής της θέσης και η κυρία Κορατσαμπίλτ με διαδέχτηκε. Πρόκειται για μια αλυσιδωτή εργασία και η έκθεση αυτή είναι απότοκη της έκθεσης της Μερέντ Μαγκίνες η οποία σας την υπέβαλε, την υπέβαλε και σε εσά και στο Προεδρείο. Πριν αναλάβω εγώ αυτό το έργο, θα ήθελα να ευχαριστήσω χαιρετήσω τη γραμματεία της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων. Χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της γραμματείας δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ανταποκριθεί, γιατί χρειάστηκε να μπορέσουμε να προοδεύσουμε σε αυτή την διαδικασία γιατί πριν ήταν μία διαδικασία διαμεσολάβησης, ενώ τώρα ε, γίνεται η εργασία μέσα στα πλαίσια ενός μεγαλύτερου συντονισμού. Ευχαριστώ λοιπόν τις δύο γραμματείς που με βοήθησαν ιδιαίτερα. Μετά από τις συστάσεις που εγκρίθηκαν από την Αντιπρόεδρο Μέρετ Μαγκίνες, ο προσανατολισμός άλλαξε τον Απρίλιο του 2018 από το Προεδρείο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο ρόλο του διαμεσολαβητή. Δεν ε, πρόκειται για μία ε, διαδικασία που ακολουθεί το, θημικό. Υπάρχει μία νομοθεσία για το ρόλο του διαμεσολαβητή. Η δική μας οργάνωση δεν ανταποκρινόταν και μετά τη συμβουλή της Μερέντ Μαγκίνες θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να εξελιχθεί αυτή η εργασία. Μιλάμε λοιπόν για τον τίτλο της συντονίστριας για τα δικαιώματα των παιδιών. Έγινε και μία ενδιαφέρουσα ακρόαση με γνωστούς επαγγελματίες που έδωσαν μεγάλη όθηση στο θέμα αυτό. Διευρύνθηκε λοιπόν η εντολή έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη την προστασία των παιδιών και την ε, πρόοδο των ε, ζητημάτων που άπτονται των διεθνών απαγωγών παιδιών. Το έγγραφο που έχετε ενώπιον σας ε, σχετίζεται με διάφορους στόχους να κάνουμε μία αποτίμηση της διετίας, να δούμε πώς εξελίχθηκε η κατάσταση από τον Απρίλιο του 2018 και ιδιαίτερα στα πλαίσια αυτής της αλυσιδωτής εργασίας να προβάλλουμε μία σειρά συστάσεων έτσι ώστε να δώσουμε μεγαλύτερο επαγγελματισμό σε αυτή την εργασία της ε, συντονίστριας. Γι' αυτό προτείνω μία συγκεκριμένη μεθοδολογία και ένα πεδίο εφαρμογής για την εργασία αυτή την οποία έχει αναλάβει η Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ τώρα, που με διαδέχτηκε πώς έχουν αυτές οι διασυνοριακές ε, γονεϊκές απαγωγές. Ε, θα ήθελα να σας μιλήσω για τη βασική δραστηριότητα που σχετίζεται και με τον ιστορικό χαρακτήρα. Ε, τι γίνεται με αυτές τις διασυνοριακές απαγωγές από τους γονείς. Δυστυχώς ακολουθούν ανωδική πορεία γιατί υπάρχει μία ε, κοινωνική συγκεκριμένη κατάσταση και παράλληλα υπάρχει δυστυχώς και ανωδική πορεία των διαζυγίων. Μετά από ε, το διαζύγιο οι γονείς πολλές φορές που προέρχονται από διαφορετικά κράτη-μέλη δεν βρίσκουν έναν κοινό τόπο για την κυδαιμονία. Και γι' αυτό το παιδί βρίσκεται είτε στη χώρα προέλευσης, είτε σε, άλλες, σε άλλη χώρα. Και πολλές φορές είναι δύσκολη αυτή η ανείχνευση των παιδιών χωρίς λοιπόν την σύμφωνη γνώμη του ενός γονέα μιλάμε για απαγωγή γιατί κατά αυτόν τον τρόπο το παιδί δεν έχει επαφή με τον ένα από τους δύο γονείς πολλές φορές χάνουμε και τα ίχνη των παιδιών. Τα παιδιά αυτά βρίσκονται στην Κεντρική Αμερική, στην Νότια Αμερική, περνάνε από μία χώρα στην άλλη και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Και γι' αυτό, μέσα στα πλαίσια της εξελικτικής πορείας, ήθελα να δράσω σε δύο επίπεδα. Καταρχήν, ως προς την πληροφόρηση των γονέων για να τους κατευθύνουμε προς ε, επαγγελματικούς κύκλους ε, που μπορούν να τους χορηγήσουν βοήθεια. Έχουμε να κάνουμε με γονείς που αντιμετωπίζουν μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα και δεν ξέρουν σε ποιο να αποτανθούν και πώς να το κάνουν. Και δυστυχώς ε, ζουν σε μια κατάσταση στέρησης Δηλαδή και τα, και τα παιδιά έχουν στερηθεί τον ένα γονέα, αλλά και ο γονέας στερείται του παιδιού του. Και γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να δράσουμε. Είμαι, ήμουν και είμαι πεπισμένη ότι θα έπρεπε αυτές τις ε, ατομικές περιπτώσεις να τις αναγάγουμε σε κάτι το πιο συλλογικό να δούμε ποια είναι τα ε, προβλήματα τα οποία ανακύπτουν συνέχεια, καθώς και τις γεωγραφικές ζώνες για να μπορέσουμε να δράσουμε και πολιτικά καθώς και διπλωματικά. Και επειδή ακριβώς έγιναν ακροάσεις στην Επιτροπή σας, με τη βοήθειά σας, είχα επαφές με τις διακοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με διάφορα φόρα που μας επιτρέπει να πλησιάσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην έκθεση αλλά θα ήθελα να τα τονίσω γιατί αφορούν μια γενικότερη τάση όπως διαγράφεται. Τα δύο αυτά χρόνια με την Βανέσα και την Ιρέν και την Στεφανή. Είχαμε 108 περιπτώσεις απαγωγής ε, παιδιών σε περίπτωση διασυνοριακών διαζυγίων ή χωρισμού. 108 περιπτώσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία αφορά ε, δύσκολες απαγωγές οι οποίες οδηγούν σε μεγάλες ρήξεις. Η ε, διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου διαρκεί χρόνια και υπάρχει και απόφαση επιστροφής του παιδιού, η οποία όμως ποτέ δεν έχει εκτελεστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνουν όλα αυτά, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση ε, στιγματισμού και στην περίπτωση που δεν γίνεται επιστροφή του παιδιού. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και πολλές φορές οι γονείς αυτοί δεν δέχτηκαν βοήθεια από τη χώρα τους και είναι, ή πρόκειται για γονείς ε, οι οποίοι ψυχολογικά και οικονομικά έχουν εξαντληθεί πλέον. Το πιο κοινό πρόβλημα είναι η μη εκτέλεση ενός ε, μίας δικαστικής εντολής σε περίπτωση επιστροφής ή οι γονείς που δεν βλέπουν το παιδί τους δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν την, ε, το δικαίωμα της επίσκεψης στο παιδί. Δεν τους επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Επίσης, στις, το 70% περιπτώσεων ε, ζήτησαν βοήθεια, ε, ζήτησε βοήθησα, βοήθεια ο πατέρας, 27% είναι οι γυναίκες, μητέρες και ένα 3% αφορά τους παππούδες του παιδιού. Το παιδί χρειάζεται τις ρίζες του για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Και αυτή είναι και η τάση παγκοσμίω που είδαμε και στη διάσκεψη της Χάγης σε σχέση με το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο. Και έτσι έχουν οριστεί και οι συνθήκες από τη δεκαετία του 80 σε σχέση με περιπτώσεις αστικού δικαίου και δίωξης δυνάμει του αστικού δικαίου. Στο 80% των περιπτώσεων η μητέρα απαγάγει το παιδί της και το μεταφέρει σε μια άλλη χώρα ή στη χώρα προέλευσής της. Στις, περιπτώσεις, στις ε, περισσότερες περιπτώσεις, ε, ως προς την κυδαιμονία ή το δικαίωμα επίσκεψης, έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο μέρος απαγωγών που ε, αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και διεθνώς. Η κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά για να αξιολογήσουμε την όλη κατάσταση και να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση. Γι' αυτό η ομάδα σας, κύριε Πρόεδρε, ασχολείται με θέματα διασυνοριακής διαμεσολάβησης και αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση αμερόληπτα. Έτσι, οι γονείς μπορούν να αποτανθούν σε επαγγελματικές οργανώσεις ε, στις οποίες έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη, δικαστές που ασχολούνται με το οικογενειακό δίκαιο, διαμεσολαβητές και ούτω καθεξής. Οι περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε παιδί δυστυχώς δεν μπορεί να έχει επαφή με την διευρυμένη οικογένεια, με έναν από τους δύο γονείς, με την γλώσσα του, τον πολιτισμό του. Πρόκειται για μία κακής μορφής ε, χειραγώγηση. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε πολιτικό επίπεδο για να μπορέσουμε να προσφεύγουμε εκεί που πρέπει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και γι' αυτό έχω κάνει και ορισμένες συστάσεις ε, μέσα στα πλαίσια της μακροχρόνιας αυτής εργασίας. Καταρχήν, διπλωματικές ενέργειες για να θίξουμε το θέμα στα κράτη-μέλη και σε τρίτες χώρες. Ε, έχω κινητοποιήσει πολλές διακοινοβουλευτικές επιτροπές, ιδιαίτερα με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και μέσα στα πλαίσια της ε, διπλωματίας και της διάσκεψης της Χάγης ε, μπορέσαμε να αλλάξουμε τους ε, διαδικαστικούς κώδικες και να βρούμε και ένα, μία δίωδο και μία διαφυγή από αυτή την κατάσταση. Το δεύτερο θέμα, ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την διεθνή οικογενειακή διαμεσολάβηση για να προωθηθεί η πρόληψη και η διαμεσολάβηση με επαγγελματικά δίκτυα, αλλά και για να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ νομικών οντοτήτων και διοικητικών δομών. Έτσι μπορέσαμε να επιλύσουμε ορισμένες δύσκολες υποθέσεις. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, έχετε την έκθεση ενώπιόν σας. Θα ήθελα να μιλήσω μόνο για τη διάσκεψη, την ε, διάσκεψη που οργανώθηκε εδώ το Νοέμβριο πέρσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είχατε ένα πάνελ επαγγελματιών που θα μας βοηθήσουν και στο μέλλον για τη διαμεσολάβηση και ακρόαση παιδιών. Και το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει ένα ζωτικό ρόλο για να βοηθήσει αυτούς τους γονείς. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για τη διαμεσολάβηση με στα πλαίσια της επίλυσης οικογενειακών διαφόρων και θα ήθελα το θεσμικό μας όργανο να κάνει ό,τι μπορεί και στην επόμενη θητεία για να προωθήσει αυτές τις ε, διαφορετικές εξοδικαστικές ε, διευθετήσεις. Εμείς συμμετέχουμε με το Ευρωπαϊκό Νομικό Δίκτυο, το οποίο συνδράμει τα κράτη-μέλη στην εργασία αυτή ως προς την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ως προς το δίκαιο των παιδιών. Πρόκειται η διευρυμένη μας ε, εντολή. Πρόκειται στο επίκεντρο να μπει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ο ρόλος του συντονιστή, της συντονίστριας. Ο ρόλος αυτός είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί και δείχνουμε αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία των δικαιωμάτων του παιδιού και δεσμεύεται στην πρόθεση αυτών των δικαιωμάτων και στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού από την πρώτη απόφαση του Προεδρείου έχουμε επεξεργαστεί τη μεθοδολογία που βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και αναπτύσσουμε ένα δίκτυο στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών επιτροπών και σε συνεργασία με όλους τους θεσμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Η συντονίστρια πρέπει να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο για όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν ε, επιπτώσεις και επηρεάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει όχι μόνο να είναι σημείο αναφορά, σημείο επαφής, αλλά κεντρικό σημείο από το οποίο απορρέει μια συνολική δράση. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι ευρωβουλευτές σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα πρέπει να μπορούμε να κινητοποιηθούμε έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε τα ψηφίσματα αυτά και όλες τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι επιμέρους βουλευτές και στα πλαίσια του συντονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι διεθνείς οργανισμοί, η κοινωνία των πολιτών, έχουν ξεκινήσει δράσεις τα δύο τελευταία χρόνια με την συντονίστρια της Επιτροπής, με την UNICEF και πολλούς άλλους οργανισμούς και ΜΚΟ. Χρειάζεται περισσότερη δράση σε επίπεδο δικτύων έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει να συνεισφέρει σε αυτή την συνολική προσπάθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι ένας δραστήριος οργανισμός, πιο αποτελεσματικός όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Φτάνουμε πολύ κοντά στις ευρωπαϊκές εκλογές και πραγματικά αυτό είναι ένας από τους ρόλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει να είναι εμφανής σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη αποστολή γιατί πρέπει κανείς να συνδυάσει ατομική δράση και συλλογική δράση, επαγγελματική δράση για πάρα πολύ ευαίσθητα λεπτά θέματα και ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε την Νομική Επιτροπή την γραμματεία σας για όλες τις προσπάθειές της τα δύο τελευταία χρόνια. Και βεβαίως ε, θα σας ακούσω με προσοχή και θα λαβώ υπόψη μου τις παρατηρήσεις σας για να υποβάλω την έκθεσή μου στο Προεδρείο. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα για ερωτήσεις από τα μέλη. Έχουμε καλέσει και μέλη της Επιτροπής Γυναικών για την σημερινή μας συζήτηση. Έχετε σχόλια, έχετε ερωτήσεις. Όχι. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν την κυρία Μωρά Σαρτιέ για όλη σας την εργασία για όλα όσα κάνετε για τους Ευρωπαίους πολίτες, για δύσκολες οικογενειακές ε, υποθέσεις. Προετοιμάζετε εξάλλου με εξαιρετικό τρόπο και την μελλοντική θητεία του συντονιστή για θέματα δικαιωμάτων του παιδιού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κληρονομιά σας είναι εξαιρετικά χρήσιμη για αυτούς που θα μας διαδεχθούν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία με την παρούσα συντονίστρια για την πρόθεση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Ελπίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τις συστάσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με την ψηφοφορία. Η πρώτη ψηφοφορία είναι για την έκθεση του κυρίου λιωτών. νομική βάση κανόνα 39, νομικές πράξεις για την ε, κανονιστική δικασία με έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια στον κύριο Λεμπριτών. Η επόμενη για την έξι της κυρίας Ρέγνερ για τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις ε, για συνοριακές ε, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Συγγνώμη κύριε που διακόπτω. Ε, αν δεχτείτε την ψήφο μου διαχειρός, επειδή περιμένουμε κάποιον να έρθει, θα σας ήμουν υπόχρεος. Άρχεται η ψηφοφορία. και λαμβάνοντας υπόψη τον κύριο Καρίμ 13 προς 2 εγκρίνεται Συγχαρητήρια στην κυρία Ρέγκνερ. Συνεχίζουμε με την εξής κυρία Ροζιέρ Θεσμικέ διαπραγματεύσει για την δράση Ευρωπαϊκή για την προσχώρηση στην πράξη τη Γενέβη, για τι ονομασίε πρόελευση και τις γεωγραφικές ενδείξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια στην κυρία Ρωσιέ. Άλλη μια έκθεση της κυρίας, της κυρίας Ροζιέρ. Σχέδιο έκθεσης. Σχέδιο σύστασης, με συγχωρείτε, για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, πράξη της Γενέβης, Συμφωνία τη Λισαβόνα για την ε, ονομασία προέλευση και τι γεωργικέ ενδείξει. Άρχεται η ψηφοφορία. και πέρας ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια κύριε Ροζιέρ. Η τελευταία ψηφοφορία για την έκθεσή μου για την αναφορά 1006 της Μπάρμπορα Στράντοβα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και για άλλη μια φορά εγκρίνεται ομόφωνα. Αυτά λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει το σημερινό πρόγραμμα. Ωστόσο, έχουμε ένα τελευταίο θέμα για την εξάδερτη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής. Θα έχουμε κοινή συνεδρίαση και ψηφοφορία μαζί με τη ΛΥΜΠΕ αύριο 2 Απριλίου και έχουμε και μια άλλη κοινή συνεδρίαση με την ΚΟΝΤ τη Δευτέρα 15 Απριλίου στο Στρασβούργο. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να τα σημειώσετε αυτά. Και θα συνθούμε στις 6 στο πέμπτο όρφο του Αλτιέρο Σπινέλη για τη συνέχιση αυτής της συνεδρίασης. Αυτή ήταν η τελευταία ανεξάρτητη συνεδρίαση. Για αυτή τη σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, την υπομονή σας. Ευχαριστώ την γραμματεία και τη βοήθεια χωρίς την οποία δεν θα μπορούσα να προεδρεύσω στην Επιτροπή. Ευχαριστώ τους διερμηνείς για το έργο τους και τη συνεισφορά τους στην επιτυχία αυτής της Επιτροπής. Και ελπίζω να ολοκληρώσουμε αυτό το εξαιρετικό έργο στην ε, συνέχεια της συνεδρίασης στις 6 ώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε ήδη, είναι η τελευταία μας συνεδρίαση ως Επιτροπή μόνη μας και το δοθείς της ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, για την εξαίρετη συνεργασία, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες και το προσωπικό της ε, ομάδας μου αλλά και την ε, γραμματεία της Επιτροπής που δεν ήταν πάντα εύκολο το έργο, το έργο της γιατί είχαμε πραγματικά πολλή δουλειά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι πάντα με χαροποιούσε ε, το να είμαι μέλος σε αυτή την επιτροπή και επειδή δεν θα ξαναέρθω αισθάνομαι ότι θα μου ξεφύγει κάποιο δάκρυ. Σας εύχομαι σε εσά που θα επανέλθετε και θέσετε στη συγκεκριμένη επιτροπή να έχετε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. πολύ δάκρυ. δάκρυ. Στις 6 ώρα λοιπόν. Σας ευχαριστώ.